θα εγκριθούν εάν ναι, αν υπάρξει αντίρρηση, θα υπάρξει πλειοψηφία. Αν έχετε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βρίσκονται στο Seance undirect. Τον Ιούλιο μετά την διακοπή, όχι, με συγχωρείτε. Τον Ιούλιο μετά την διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού μας συνυπέγραψα με τον πρόεδρο του Συμβουλίου τρεις νομοθετικές πράξεις. Θα υπογράψω και αυτή την εβδομάδα περαιτέρω νομοθετικές πράξεις. Οι τίτλοι ε, των υπογεγραμμένων πράξεων και αυτών οι οποίες θα υπογραφούν θα δημοσιευτούν με τα πρακτικά αυτή τη συνεδρίαση. Περνάμε τώρα στην υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τη μορφή που έχει. Έχω μόνο μία